μία προφορική ερώτηση προς την Κομισιόν εφαρμογή του άρθρου 20 παράγραφος 2 της οδηγίας για τις υπηρεσίες και του άρθρου 8 παράγραφος 3 της οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Θα δώσω τώρα τον λόγο σε αυτούς οι οποίοι έκαναν την ερώτηση στην κυρία Γκέπχαρτ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ, εδώ είμαι. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας ε, δίνεται να κάνουμε αυτή την ερώτηση. Διαπιστώνουμε πως όλο και συχνότερα οι πολίτες κάνουν αγορές στο ίντερνετ και για διάφορους λόγους ε, δεν μπορούν να το κάνουν αυτό γιατί έχουν λάθος διεύθυνση IP, έχουν λάθος ε, πιστοτική κάρτα, ζουν σε λάθος χώρα, έχουν λάθος υπηκοότητα και άρα δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν μια συναλλαγή. Το δίκαιο όμως εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ξεκάθαρο. Διακρίσεις λόγω ηθαγένειας ή τόπου κατοικίας δεν είναι αποδεκτή. Οπότε είναι απαράδεκτο σήμερα σε αυτή τη μεγάλη εσωτερική αγορά που έχουμε, που είναι πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για τις επιχειρήσεις, να μην υπάρχει τελικά για τους καταναλωτές και να υπάρχουν όλα αυτά τα εμπόδια. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να κάνουμε κάτι. Και στην ε, ανακοίνωσή σας για την ε, στρατηγική, για μια ψηφιακή εσωτερική αγορά για την Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναφέρω επιλέξη είπε για το 2016 θα σταματήσει το αδικαιολόγητο γεω... τον αδικαιολόγητο γεωγραφικό αποκλεισμό στην περίπτωση ηλεκτρονικών συναλλαγών. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω τι εννοείται με αυτή την αλλαγή, τι μορφή θα έχει και τι στόχο έχετε εδώ πέρα. Επίσης με ενδιαφέρει πάρα πολύ να γνωρίζω τι σκοπεύετε να κάνετε για την ορθή εφαρμογή του άρθρου 22 και του άρθρου 8.3 των οδηγιών για τις υπηρεσίες και τις προστασίες των καταναλωτών. Δικαιώματα τα οποία υποτίθεται πως υπάρχουν, αλλά εξακολουθούν να μην ισχύουν για τους πολίτες. Θέλω λοιπόν να ακούσω τι θα μας πείτε. Σας ευχαριστώ. Σβάμπ για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σημερινή προφορική ερώτηση προς την Κομισιόν μας δίνει την ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε ακόμη μια φορά το τι θέλουμε και το τι ορίσαμε ως νομοθέτες στις δύο αυτές ε, οδηγίες. Η άνηση μεταχείριση καταναλωτών με βάση εθνικότητα ή τόπου κατοικίας επιτρέπονται μόνο εάν υπάρχουν ουσιαστικοί νόμιμοι λόγοι. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμείς προσπαθούμε ακριβώς να δημιουργηθούν οι κατάλληλες ε, προϋποθέσεις για να μην είναι δυνατόν πλέον να υπάρχει διαφορετική μεταχείριση. Ξέρουμε πως χρειάζεται να γίνουν κάποια πράγματα έτσι ώστε οι επιχειρήσεις αφενός και οι καταναλωτές αφετέρου πραγματικά να έχουν ένα ενιαίο περιβάλλον. Αυτό το οποίο βλέπουμε όμως σε κάποιες επιχειρήσεις, θα αναφέρω την επιχείρηση Disneyland ε, το καλοκαίρι, παρά το ότι λοιπόν υπάρχουν οι συνθήκες υπάρχει μια προσπάθεια να ε, βάλουν διαφορετικές τιμές ανάλογα με το από πού προέρχεται κανείς στην Ευρώπη. Και αυτό είναι πραγματικά απαράδεκτο. Πρέπει λοιπόν η Κομισιόν να κινητοποιηθεί με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της. Και αυτό το λέω γιατί γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι να είναι ενιαίες οι συνθήκες. Έχουμε πάντα τη συζήτηση για το πώς ενιαία μεταχείριση μπορούμε να αντέξουμε. Υπάρχουν κράτη-μέλη που δεν θέλουν εναρμόνιση των νομικών συνθήκων, αλλά ακόμα και εκεί όπου υπάρχει νομική εναρμόνιση, τελικά ο καταναλωτής λαμβάνει την εντύπωση πως ε, οι επιχειρήσεις καρπώνονται τα ωφέλη της ενιαίας ε, αγοράς, αλλά μετά δεν κάνουν τίποτα για τον καταναλωτή. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω κύριε Επίτροπε, τι θα κάνετε εδώ πέρα. Σας ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Γιάκοφτιτς. Ευχαριστώ. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά υπάρχει πρόβλημα με την κροατική διερμηνία. Πριν δεν ακούσαμε τα γερμανικά, μετά τα αγγλικά. Υπάρχει πρόβλημα με την κροατική ε, διερμηνία. Προσπαθώ να καταλάβω, αλλά δεν μπορώ να τα καταλάβω όλα. Παρακαλώ φροντίστε να αποκατασταθεί η κροατική διερμηνία. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε. Ναι, θα φροντίσουμε να ενημερωθούν ε, οι τεχνικές υπηρεσίες. Μας το είπατε και προηγουμένως. Κύριε Επίτροπε, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Με συγχωρείτε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκ μέρους της ε, συναδέλφου Εκ μέρου του συναδέλφου λοιπόν της Αρμόδιας Επιτρόπου πρέπει να πω ότι το θέμα που θέτουν ε, οι βουλευτές αγγίζει πραγματικά την ουσία των προσδοκιών των πολιτών από την ενιαία αγορά. Αγορές διασυνοριακές. Όμως στη διακριτική μεταχείριση υπάρχει βάση της υπηκότητας ή του τόπου κατοικίας και αυτό είναι απαράδεκτο σε μια ενιαία αγορά. Διαρκώς λαμβάνουμε παράπονα και προσφυγές ε, από τους πολίτες για τις ε, αθέμητες πρακτικές ε, ίσο κάποιες φορές άμεσες προσφυγές στα, καταναλωτικά, στα κέντρα για τους Ευρωπαίους καταναλωτές και έπειτα πολλές φορές και αιτήσει για την παροχή συμβουλών και κοινοβουλευτικές ερωτήσεις σε κάποιες περιπτώσεις. Ως δημοκρατικά εκλεγμένοι εκπρόσωποι των πολιτών είστε πραγματικά ο σημαντικότερος συνομιλητής μεταξύ των πολιτών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Ε, βεβαίως, ε, καλά κάνετε και μας ενημερώνετε το συμβαίνει στις εκλογικές σας περιφέρειες. Η εφαρμογή των κανόνων του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι σημαντικότατη, αλλά ε, πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι κανόνες για τις ηλεκτρονικές ε, συναλλαγές. Ο γεωγραφικός αποκλεισμός είναι ένα από τα βασικά είδη ε, διακριτικής μεταχείρισης που εντοπίζουν οι καταναλωτές στις διασυνοριακές συναλλαγές τους. Η αγορά τους μπλοκάρεται ή επανακατευθύνονται σε ένα νέο ιστότοπο για την παροχή της ίδιας υπηρεσίας αγαθού, αλλά με υψηλότερη τιμή. Η διακριτική μεταχείριση μεταχείριση ασκείται σε καθημερινή βάση ει βάρο εκατομμυρίων Ευρωπαίων που ταξιδεύουν στο εξωτερικό ω τουρίστε και αγοράζουν μια δευτερεύουσα ε, κατοικία, ένα σπίτι λοιπόν ε, ε, σε άλλη χώρα ή απλώς διασχίζουν τα σύνορα. Αυτό πρέπει να πάυσει στα πλαίσια και τη ενιαίας ψηφιακή αγοράς. υπάρχει ανάγκη για δράση και θα πρέπει αυτό το να καλύψει και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές για την πόλη και αγορά ε, αγαθών και υπηρεσιών διαδικτυακά. Ήδη ξεκινήσαμε δημόσιες διαβουλεύσεις ε, για να μπορέσουμε να προκάνουμε μια νομοθετική πρόταση εντός της επόμενης χρονιάς. Ξέρουμε πόσα παραδείγματα διαγετικών ε, πρακτικών μπορεί να παριθμίσει κανείς. Πέρυσι ξεκινήσαμε μία ε, διαδικασία μελέτης για να δούμε τι γίνεται με τις εταιρείες σας αυτοκινήτων ε, ανά την Ευρώπη και να δούμε γιατί υπάρχουν τέτοιες διαφορετικές τιμές ανάλογα με τον τόπο κατοικίας του πελάτη. Φέτος Είδαμε τι γίνεται με ένα μεγάλο κέντρο ψυχαγωγίας ε, στην ε, Γαλλία, ένα, Luna Park, ένα είδος Λούνα Πάρκ που πολλές φορές περιορίζεται μόνο στους ε, ντόπιου, σε Γάλλους. Επίσης ξέρουμε τι γίνεται με τους ε, πελάτες που χρειάζεται να έχουν έναν, ε, ε, ένα αριθμό φορολογικού μητρώου σε κάποιες χώρες για να κάνουν μια συγκεκριμένη αγορά. Ε, πρέπει αυτό να δούμε ότι δυσκολεύει και τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές και δεν επιτρέπει τις αθηνικές αρχές να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για την ίδια και μεταχείριση σε καθημερινή βάση. Αυτό θέλουμε να αντιμετωπίσουμε. Η συμβασιακή ελευθερία είναι μια θεμελιώδης αξία που πρέπει να διαφυλαχθεί. Αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τον δευτερογενή κατακαιρματισμό της ενής αγοράς από εταιρείες που διαρκώς ε, καταπατούν τα δικαιώματα των καταναλωτών. Οι ανάγκε των μικρομεσαίων επιχειρήσεων πρέπει επίση να καλυφθούν. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τι εταιρείε και του καταναλωτέ να ε, ε, αξιοποιήσουν την ενιαία αγορά προ όφελό του. Δεν θέλουμε να υπάρχει αβεβαιότητα. Ε, συνάδελφοι, κυρία Μπιάνκοφσκα και ο κύριος Τιγκέρ με τα χαρά θα συζητήσουν τις αναγκαίες αλλαγές προκειμένου να βελτιωθεί η νέα αγορά όπως διατίθεται στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Ευχαριστούμε. Να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Σενάλοβα για να Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η διάκριση βάρος των καταναλωτών εξαιτίας της του τόπου διαμονής ή ε, της ε, εθνικότητάς τους είναι πραγματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλιστεί μια ασφάλεια δικαίου με αντικειμενικά κριτήρια και με καθορισμό των προϋποθέσεων ε, και μόνο με εξαιρετικές, σε εξαιρετικές περιπτώσεις να υπάρχει περιορισμό στην πρόσβαση αγαθών και υπηρεσιών. Επίσης, οι αρχές ελέγχου θα πρέπει να διενεργούν καλύτερα τον έλεγχο για να πεταχθεί αυτή η διάκριση εις βάρος καταναλωτών. Βέβαια, η εξάλληψη αυτού το προβλήματος είναι από τις σημαντικότερες προκλήσεις της εσωτερικής αγοράς. Οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν διακρίσεις ε, και στο διαδίκτυο αλλά και εκτός του διαδικτύου. Θα πρέπει να μην υπάρχουν διαφορές, να μην υπάρχουν αντιφατικές διατάξεις ε, για τις πωλήσει on και offline. Ελπίζω να συνεχίσει τις προσπάθειές της Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να εφαρμόσει το σχέδιο δράσης. Η κυρία Χαράνζοβα, παρακαλώ, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει μάχη για το θέμα αυτό και οι φιλελεύθεροι ε, ελπίζουν ε, να υιοθετηθεί η οδηγία αυτή για το geo-blocking και να καταλαμβάνει και τις οδηγίες για τις υπηρεσίες και τα αγαθά. Είναι δύσκολη η αγορά διασυνοριακά για τους καταναλωτές, γιατί μερικές φορές ε, δεν μπορούν να λάβουν τα αγαθά τους. Ε, η παράδοση είναι τόσο δαπανηρή που τελικά δεν φτάνουν τα αγαθά στον καταναλωτή. Αν τα αγαθά και το περιεχόμενο δεν μπορεί να περάσει τα σύνορα, τότε προστεί διασυνοριακέ αγορέ. Θα μένουν περίκλειστοι και εγκλωβισμένοι στι εθνικέ αγορέ οι καταναλωτέ και θα υφίστανται υψηλότερε τιμέ εξαιτία τη έλλειψη πλήρου και θεμητού ανταγωνισμού. Κύριε Επίτροπε, ε, αν το συγκρίνουμε και με τις διαφορετικές τιμές ανάλογα με τον τόπο πώλησης, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει κατάφορη ε, διάκριση ε, εις βάρος των καταναλωτών από πλευράς επιχειρήσεων. Ε, διάκριση είτε λόγω εθνικότητας είτε λόγω τόπου διαμονής. Όχι γιατί είμαι Τσέχος, αλλά γιατί ζω στην Πράγα. Μερικοί λένε ότι δεν ισχύει διάκριση αλλά απλώ ε, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το θέμα των επιστροφών ή το γλωσσικό ζήτημα. σω έχουν δίκιο οι επιχειρήσει. σω θα πρέπει να επικεντρωθούμε και σε αυτά τα προβλήματα, όπω προβλέπεται άλλωστε και στη στρατηγική. Όμω, κύριε Επίτροπε, με τι, λόγο, με τι λόγους ε, μία πολυεθνική μπορεί να δικαιολογήσει αυτή την άρνηση παροχής υπηρεσιών. Γενικώ είμαι κατά τη υπερβολικής ρύθμιση ε, για τις επιχειρήσεις, αλλά ειλικρινά πιστεύω ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι καλοπροαίρετες και θέλουν να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους και να αυξήσουν και την πελατεία τους. Αλλά εδώ έχουμε μια περίτρανη απόδειξη και κατάφορη περίπτωση που απαιτεί δράση για να ε, καταπολεμήσουμε τη διάκριση και τον κατακαιρματισμό της αγοράς. Πρόκειται για σαφή διάκριση των τιμών, που είναι απαράδεκτη σε μια ενιαία ψηφιακή αγορά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο κύριος Σοφλίν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία όλα αυτά. Η Κομισιόν τονίζει το πρόβλημα του γεωγραφικού αποκλεισμού και παριστάνει τον υπερασπιστή του καταναλωτή, αλλά και η Κομισιόν είναι ο πρώτος γεωγραφικός αποκλειστής καθώς έχει κάνει πάρα πολύ δύσκολο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, το να πουλάνε στο εξωτερικό. Με τελευταίο χαρακτηριστικό παράδειγμα φόρο ηλεκτρονικού εμπορίου σε κάθε χώρα στην οποία πουλάνε. Οπότε δεν εξάγουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μικραίνουν οι επιλογές των καταναλωτών. Πάρα πολύ συχνά λοιπόν η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το πρόβλημα και όχι η λύση. Ε, δεν αφιβάλλω ότι έχετε καλές προθέσεις, αλλά πρέπει να δείτε το τι κακό κάνετε στην πράξη. Στην Ήπειρο, η οποία πλέον θα γίνει η λιγότερο οικονομικά δυναμική του κόσμου. Σας ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στη διαδικασία Catch Τέσσερις συνάδελφοι θα πάρουν το λόγο. Ο κύριος Καπούτο. Η κυρία Γκραπίνη, γιατί δεν βρίσκεται στην αίθουσα ο κύριος Καπούτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ξεκινήσω συγχαίροντας τους συντάκτε της προφορικής ερώτησης. Συμμετέχω στην Επιτροπή Προστασίας των Καταναλωτών και το θέμα αυτό το συζητούμε συχνά. Δεν αρκεί η οδηγία για τις υπηρεσίες, εάν δεν παρακολουθούμε σωστά τι συμβαίνει στην αγορά, βεβαίω θέλουμε ένα νέο πλαίσιο. Και όπως σωστά υπόθηκε, κάποιες φορές αναγκάζεται κανείς να πάει σε άλλη χώρα για να αγοράσει κάτι στο διαδίκτυο. Επίσης το κόστος της παράδοσης, οι καθυστερήσεις και άλλα σχετικά ζητήματα. Νομίζω ότι σημαντικό είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη αυτές τις ε, προσδοκίες. Περιμένω όμως και μια συγκεκριμένη απάντηση. Τι θα κάνουμε για να βελτιώσουμε την ποιότητα, για να επιβάλλουμε με τρόπο ομοιόμορφο την οδηγία για την παροχή υπηρεσιών σε όλες τις χώρες και να αποφύγουμε κάθε είδους διακριτική μεταχείριση. Πρέπει να δράσουμε εγκαίρως και ε, στο επίπεδο της πρόληψης, όχι των Συζητούμε για τα δικαιώματα των καταναλωτών και πώς τα κράτη-μέλη θα πρέπει να φροντίσουν ώστε να μην γίνονται διακρίσεις λόγω ηθαγένεια και τόπου κατοικία που παραλείπει. αρχικά τα κράτη μέλη οφείλουν να επιβλέπουν τη σωστή εφαρμογή τη υπάρχουσα νομοθεσία, όσον αφορά τι διαδικτυακέ υπηρεσίε. συχνά ορισμένοι καταναλωτέ, προερχόμενοι από μικρά κράτη μέλη έρχονται αντιμέτωποι με αρκετέ δυσκολίε κατά τη διαδικασία παραλαβή των αντικειμένων που επιθυμούν ενώ σε ορισμένε περιπτώσει, οι διαδικτυακέ υπηρεσίε αρνούνται να παραδώσουν τα αντικείμενα στου καταναλωτέ είναι επομένως αναγκαίο η ευρωπαϊκή ένωση να βάλει τέλος στον αδικαιολόγητο αποκλεισμό των καταναλωτών από την αγορά οποιονδήποτε αγαθών ή υπηρεσιών εφόσον αυτή η κίνηση παραβιάζει τα βασικά τους δικαιώματα. επιπλέον στα πλαίσια του ηλεκτρονικού εμπορίου θα πρέπει να σταματήσει η επιπλέον επιβάρυνση του καταναλωτή για το κόστος μεταφοράς σε περίπτωση που δεν έχει ενημερωθεί από πριν γι' αυτό. Τέλος, θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα από την ευρωπαϊκή ένωση ώστε να υπάρξει μια στοχευμένη αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής του ηλεκτρονικού εμπορίου χωρίς να καταπατώνται τα δικαιώματα των καταναλωτών. ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ε, ο γεωγραφικός αποκλεισμός, το geo-blocking, είναι από τις πιο ύπουλες διακρίσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα στην ε, ψηφιακή αγορά. Και είναι από τα σημαντικότερα εμπόδια των νέων τεχνολογιών ε, που εμποδίζουν τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Εμείς είμαστε υπέρ της ενιαίας ψηφιακής αγοράς ε, και σήμερα αντιμετωπίζουμε εμπόδια από την ίδια τη τεχνολογία που μας εμποδίζει να προχωρήσουμε και από προσωπικές ε, εμπειρίες που είχα, αλλά και από εμπειρίες συναδέλφων, θα ήθελα να απευθύνω έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει ό,τι μπορεί, να μην φυστεί προσπαθειών και όσο το δυνατό γρηγορότερα να πατάξει αυτό τον ύπουλο τρόπο διάκρισης που είναι ο γεωγραφικός αποκλεισμός. Μόνο έτσι θα αναπτύξουμε μια πραγματικά ενιαία ψηφιακή αγορά. Σας ευχαριστώ. Κύριο Καπούτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η δημιουργία της ψηφιακής πώληση αγαθών ε, και των διασυνοριακών συναλλαγών είναι σημαντικές για να ξεπεράσουμε τα εθνικά σύνορα και να εφαρμόσουμε την ε, ενιαία ψηφιακή αγορά στην Ευρώπη. Όμως η προστασία των καταναλωτών ε, πρέπει να είναι μια υψηλή προτεραιότητα ώστε να υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο προστασία και για τις συναλλαγές και για την απόκτηση των επιθυμητών αγαθών χωρίς το γεωγραφικό αποκλεισμό. Θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στις διαδικασίες αγοράς επιγραμμικά με ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο και ισότητα στην παροχή υπηρεσιών. Δεν μπορούμε να παραβλέπουμε τα δείγματα που έρχονται από την τελευταία αποφάση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 6 ε, Οκτωβρίου του 2015 που καθορίζει ότι η, παροχή ευαίσθητων πληροφοριών από τα προσωπικά δεδομένα του ε, καταναλωτή πρέπει να είναι κάτι που να λαμβάνεται υπόψη και να μην υπάρχει η διακριτική μεταχειρίση βάσει του γεωγραφικού αποκλεισμού. Θα πρέπει να ληφθεί λοιπόν αυτή η απόφαση υπόψη, να δημιουργήσουμε ένα πραγματικό ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο για την ενιαία ψηφιακή αγορά και να προτεύουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών ανεξαρτήτω ηθαγένεια. Ευχαριστούμε. Έχετε το λόγο κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ Πρόεδρε να σας ευχαριστήσω και πάλι για τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα για την προστασία των καταναλωτών και τις διακρίσεις εναντίον τους. Εδώ μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι η τρέχουσα κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Υποσχόμαστε στους πολίτες να είναι καταναλωτές εσωτερικής αγοράς με την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί υποτίθεται ότι έχουμε πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες και την ηλεκτρονική αγοραπολισία αγαθών. Και όμως πολλές φορές αυτό δεν ισχύει, διότι τα προσφερόμενα δεν ε, προσφέρονται σε μια συγκεκριμένη χώρα ή δεν υπάρχει ίση δίκαιη μεταχείριση σε σχέση με τον καταναλωτή μιας διαφορετικής χώρας. Η εσωτερική αγορά σημαίνει ίδια προσφορά προς όλους με ίδια πρόσβαση, ίση πρόσβαση από οποιοδήποτε σημείο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο καθένα θα πρέπει να μπορεί να αποκτήσει ό,τι επιθυμεί ακόμη και από άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Να είμαι σαφή. Οι ελευθερίε πάντοτε πρέπει να αντισταθμίζονται με κάποιες άλλες. Δεν είναι κανείς σημαντικότερος κάποιου άλλου. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε συμβασιακή ελευθερία και οι καταναλωτές να μην πέφτουν θύματα διακρίσεων λόγω του τόπου κατοικίας τους. Επίσης θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν υπάρχει υποχρέωση να ενοποιήσουμε τις τιμές μέσω της ενιαίας αγοράς το ποιο είναι το σωστό σημείο ισορροπίας θα εξαρτηθεί και από το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων και τις συζητήσεις με τους ενδιαφερομένους στα κράτη-μέλη. Το άρθρο 20 της υπηρεσίας για τις οδηγίες καθορίζει τις ε, υποκείμενες, τις βασικές αρχές που θα πρέπει να ε, μεταφέρουν και να εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη. Αν κάποιο κράτος παραβιάζει την αρχή αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να εκινήσει τη διαδικασία παραβάση εναντίον του. Ε, φαίνεται ότι πολλά κρατημέλη δεν έχουν ε, αναλάβει αρκετέ δράσει, ώστε η αρχή τη μη διακριτική μεταχείριση να εφαρμοστεί. Οι διαδικτυακέ αγορέ έχουν επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα για τη δημιουργία ενό συνεκτικότερου, πιο ε, ενιαίου, ομοιόμορφου και φιλικού προ τον καταναλωτή πλαισίου. Θα γίνουν λοιπόν οι ανάλογε προτάσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την παρουσίαση τη στρατηγική για την ενιαία ε, ψηφιακή αγορά και το ενιαίο θεματολόγιο. Ευχαριστούμε κυρία Πίτροπε. Κλείνει η συζήτηση για το θέμα αυτό και περνάμε στο επόμενο.